της συνεδρίασής μας συνεχίζεται η Ολομέλεια αύριο το πρωί στις 8.30 μέχρι τις 2 και μετά από τις 3 μέχρι τις 11.